να είναι και σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με την Πολωνία γιατί ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι θέμα και των θεσμών αλλά και των κρατών μελών. Είναι ένα ουσιώδες κομμάτι της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και είναι η βάση για την εμβέα εμπιστοσύνη και την αναγνώριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγική επεξήγηση της κατάστασης. Ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μέλλον για το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Ε, ξεκινάμε με την ε, κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, τον κύκλο των πολιτικών ομάδων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ενδεικτικό τη κατεπίγουσα κατάσταση το γεγονό ότι σήμερα πάλι συζητούμε για την Πολωνία. Βρισκόμαστε εδώ γιατί και οι Πολωνοί πολίτε είναι Ευρωπαίοι πολίτε και αξίζουν την ίδια προστασία και τα ίδια δικαιώματα με του πολίτε τη Σουηδία, τη Ιταλία ή τη Γερμανία. Και θα πρέπει να έχουν δυνατότητα προσφυγή στη δικαστική εξουσία. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πρόσβαση. Έχουν μπλοκαριστεί όλε οι διέξοδοι προ τη δικαστική εξουσία. Γι' αυτό και καλούμαστε να λάβουμε το ρόλο μα. Είμαστε εδώ έσχατο μέσο και έκκληση προς την πολωνική κυβέρνηση διαρρέξει το διάλογο και όχι την αντιπαράθεση, ε, την δικαιοσύνη και όχι την προκατάληψη. Και είναι ηρωνικό πραγματικά που την τελευταία φορά που είχαμε τέτοια πίεση της κυβέρνησης ε, στη δικαστική εξουσία ήταν πριν το 1989. Και αυτό που έκανε ουσιαστικά η σημερινή πολωνική κυβέρνηση είναι να παλινδρομήσει προς το παρελθόν. Χρησιμοποίησε αυτή την επαναχώρηση και την καταπίεση που αντίκειται σε οποιαδήποτε αξία και αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό δώσαμε τον αγώνα μας, γι' αυτό πολεμήσαμε, για να καταργηθεί τέτοια καταπίεση. Πάντως, οι γενναίοι Πολωνοί δικαστές το αντίθετο διεκδικούν και με τιμή και σεβασμό αντιμετωπίζουμε τους Πολωνούς δικαστές γιατί το θάρρος τους και ο όρκος τους είναι σύμβολο του πολωνικού κουράγιου που ο κόσμος θαυμάζει θα υπάρξουν συνέπειε με την καταστρατήγηση του δικαίου. Υπάρχουν κανόνε που όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να εφαρμόσουν εφόσον εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν αμέσω να εφαρμοστούν ε, ε πρόσωρινα μέτρα για να αποφευθεί η καταπίεση και να προστατευτεί ο ευρωπαϊκό τρόπο ε, και οι Πολωνοί πολίτε. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει η Πολωνία να εκτραπεί προς τέτοια αυθαιρεσία. Ε, εμείς ε, ε, λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, και τη Βολωνική Κυβέρνηση να μην γυρίσουν την πλάτη τους στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο συνάδελφος Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε Γιώργο, όπως ξέρετε, έχω την τιμή να προεδρεύω στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, που συζητά ακριβώς ε, την τήρηση των αρχών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, το, τις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, που δεν είναι ο κανόνας της ε, πλειοψηφίας, αλλά ο σεβασμός της μειοψηφίας και υπάρχει δικαίωμα στην αντιπολίτευση, δικαίωμα στον ε, αντίλογο και φυσικά προστασία της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας. Θα πρέπει λοιπόν να, να εφαρμόσουμε ε, το άρθρο 7 και για την Ουγγαρία και πάλι να το εφαρμόσουμε και για την Πολωνία που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Γιατί είχαμε μια συσσόρευση νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στην Πολωνία που απειλούν σοβαρά την ανεξαρτησία του, της δικαστικής Το πειθαρχικό τμήμα που ε, από το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κηρύχθηκε ε, αντίθετο με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η απειλή επιβολής κυρώσεων προς τους δικαστές που διαφωνούν είναι απαράδεκτα. Και Γι' αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε την αμέριστη υποστήριξή μας προς προνούς δικαστές. Θα πρέπει να φέρετε εις πέρας την εντολή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, κύριε Αντιπρόεδρε, Υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου που θα πρέπει να είναι αντικειμενικός μόνιμος, ε, να συμπεριλαμβάνει τους πάντες, να μην έχει αποκλεισμού και με περιοδικό τρόπο να εξετάζει την εφαρμογή των αρχών του ενωσιακού δικαίου και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέπουμε κάτι που χαρακτηρίστηκε ως συνταγματική ε, ανατροπή, ως ε, ουσιαστικά αντισυνταγματική συμπεριφορά και παλιδρόμηση της Πολωνίας προς μια ε, κατάσταση αντίθετη με το νοσιακό δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον συνάδελφο Σίμισκα από την ομάδα Renew Europe. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, Αγαπητέ, Επίτρο, αγαπητή Επίτροπε, θυμάμαι πριν από τέσσερις εβδομάδες είχαμε την ε, συζήτηση αυτή και θυμάμαι που είχα πει ότι η κατάσταση στην Πολωνία είναι άνευ προηγουμένου. Ουδέποτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαμε κυβέρνηση κράτους μέλους που να ασκεί τόσο έλεγχο στη δικαστική εξουσία. Και τέσσερις εβδομάδες μετά, ένα μήνα μετά, βρισκόμαστε και πάλι να συζητούμε το ίδιο θέμα με την κατάσταση να έχει επιδεινωθεί. Ε, η Πολωνία είναι το πρώτο κράτος μέλος που εφαρμόζεται στο νοσιακό δίκαιο. Παρόλα αυτά ε, ε, μπορεί να απολύσει δικαστές. Ε, ουσιαστικά ασκεί έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας στις υποτιθέμενα ανεξάρτητους δικαστές. Και μάλιστα το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο φαίνεται ότι είναι όμοιρος αυτής της κατάστασης ε, και έχει καταργηθεί διάκριση εξουσιών σε ένα κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει, όχι για να τιμωρήσει την Πολωνία ή την πολωνική κυβέρνηση, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να δράσουμε για να προστατεύσουμε τα πολιτικά και δημοκρατικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, Εν προκειμένου των Πολωνών πολιτών. Και ακούσαμε ότι υπάρχει μια προκατάληψη εις βάρος Πολωνίας αυτό ισχυρίζονται οι κυβερνώντες ότι δεν καταλαβαίνει η Δύση τι σημαίνει η παρακαταθήκη του κομμουνιστικού καθεστώτος και όμως ε, Είμαι πολιτικός ε, ε, και η οικογένειά μου έχει διωχθεί από την κομμουνιστική ε, δικαστική εξουσία και δεν έχει καμία θέμα, κανένα θέμα αυτό με την νομική παράδοση ενός κράτους, αλλά με την υποστήριξη των δικαστικών παραδόσεων και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον Σάλφα Μπλάσκο από την ομάδα ID. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο είναι αξιοπρόσεκτο. Το γεγονός ότι για άλλη μια φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούμε μια δήλωση που αφορά στο απειλούμενο κράτος δικαίου στην Πολωνία. Συζητούσαμε πριν γιατί έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα έπρεπε μάλλον να συζητάμε και αυτή τη φορά. Ε, αλλά για άλλη μια φορά συζητάμε την Πολωνία για το πώς ε, ε, ο η εθνική κυριαρχία και ο πατριωτισμός ε, γίνονται θέμα σε μια χώρα όπως η Πολωνία. Έχουμε λοιπόν την καθημερινή ζωή πολιτών ε, που ετίθεται ε, υπό αμφισβήτηση και ακούμε αιτιάσεις σχετικά με μια εκστρατεία κατά της Πολωνίας η οποία θέλει να θεσπίσει τη δική της μορφή δημοκρατίας. Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να επεμβαίνει στα εσωτερικά ενός κράτους μέλους. Όποτε έχει συμβεί αυτό στην ιστορία δεν ήταν σωστό. Σας ζητώ. Αυτό γιατί το κάνετε λοιπόν, για να έχουμε ένα αντόμινο. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Ράντκε για τους πράσινους παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Ένα πράγμα ισχύει. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να χτίσεις ένα δημοκρατικό σύστημα, ούτε και οι νομικές παραδόσεις ε, στην Ευρώπη είναι ίδιες. Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση για όλα τα καταστάσεις. Το να έχεις πλειοψηφία δεν σημαίνει ότι μπορείς να υποσκάπτεις το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και το λέω αυτό γιατί και τα δύο είναι αυτή τη στιγμή δέχονται επίθεση στην Πολωνία. Η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος ε, ο διαχωρισμό των εξουσιών, όλα αυτά είναι σημαντικά και δέχονται επίθεση. Υπάρχει ο νόμο του πιο ισχυρού και παίρνουμε δικαιώματα από αυτού που είναι εύκολο να του τα πάρουμε. Στο μέλλον λοιπόν η συζήτηση για το άρθρο 7, ο μηχανισμό για το κράτο δικαίου, η μελλοντική συζήτηση, όλα αυτά θα πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη του ε, στη μελλοντική συζήτηση που θα γίνει. Χωρί την Πολωνία η Ένωση δεν μπορεί να είναι ποτέ ολοκληρωμένη γιατί οι Πολωνοί πολίτε είναι όντω Ευρωπαίοι πολίτε. Αντί λοιπόν να, ε, να κατηγορούμε τι Βρυξέλλε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή οποιονδήποτε θέλουμε για αυτό που συμβαίνει, καλό θα ήταν η πολωνική κυβέρνηση να ξεκινήσει έναν ανοιχτό επικοδομητικό διάλογο για να επιληθεί αυτό το επίπεδο πήγον και σημαντικό πρόβλημα και σας καλώ συναδελφοί να φέρετε αυτό το μήνυμα στην Πολωνία. Και όπου και αν βρίσκεστε εδώ στο φάσμα αυτής της συζήτησης, ε, όποια και εκστρατεία και αν έχετε ακολουθήσει στο περασμένο μήνα, τα περασμένα χρόνια, το, είχαμε πολλές περιπτώσεις που μιλήσαμε για την Πολωνία. Είναι αν παράδεκτο. Δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατική συζήτηση αν δεν σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είδα μια μπλε κάρτα, αλλά συνήθως δεν έχουμε μπλε κάρτες στον πρώτο γύρο για τις ομάδες, οπότε αν θέλετε μπορείτε να τη δεχτείτε αργότερα. Όχι στον πρώτο γύρο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον συνάδελφο Τσίτλο εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, η Πολωνία είναι υπέρ της ενίσχυσης του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό τον όρο όμως ότι θα εθράζονται στη συνθήκη και δεν θα επηρεάζουν την ε, εθνική ταυτότητα των κρατών μελών. Θα έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα και δεν θα επιβάλλουν διακρίσεις εις βάρος μερικών κρατών μελών. Κρίμα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί ε, μια πολιτικοποιημένη κατάσταση και ε, εργαλειοποιεί το θέμα του κράτους δικαίου. Το πολωνικό σύστημα δικαιοσύνης απαιτεί μεταρρυθμίσεις. Εδώ και τέσσερα χρόνια η πολωνική κυβέρνηση με βάση το πολωνικό σύνταγμα και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται και από τη συνθήκη και ανάλογα με τις προσδοκίες των πολωνών πολιτών που είναι η κυρίαρχή μας ε, διεξαγάγει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ξεκινήσαμε τη μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας και αυτή τη μεταρρύθμιση θα την ολοκληρώσουμε είναι γεγονός ότι στην ε, Πολωνία έχουμε μια πολιτική διένεξη, αλλά θα αποφανθούν τα πολωνικά δικαστήρια και, και σίγουρα ε, αυτό είναι αρμοδιότητα της Πολωνίας και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η παρεμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτά είναι που καταστρατηγούν τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Ε, δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς για τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, της δικαστικής εξουσίας στη Γαλλία ή την, το διορισμό των δικαστών από το Κοινοβούλιο στη Τσεχία ή σε άλλη χώρα. Οπότε δεν είναι μόνο κατάσταση της μεταρρύθμισης αυτής πολωνικό χαρακτηριστικό. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε την μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας και με βάση τη συνθήκη τη συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χώρα μέλο έχει δικαίωμα να κάνει τέτοιε μεταρρυθμίσει. Η σημερινή συζήτηση έχει πολιτική διάσταση και είναι τελείω ανεδαφική και δεν ε, στηρίζεται σε κανένα πραγματικό ε, λόγο παρά μόνο στην, στα πολιτικά κίνητρα. Στην Πολωνία σας διαβεβαιώ ότι έχουμε κράτος δικαίου και δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε αυτό το θέμα για την Πολωνία. Ε, δημιουργείται μια εικονική εντύπωση για την Πολωνία. Δεν ισχύει αυτό. Η Πολωνία σίγουρα είναι έτοιμη για διάλογο και συνεργασία. Αλλά για να είναι εφικτή ε, αυτά ο διάλογος και η συνεργασία θα πρέπει να υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές και όχι μόνο από την πολωνική πλευρά. Εδώ και τέσσερα χρόνια ξεκινήσαμε μεταρρυθμίσεις που σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί λοιπόν σας ενοχλούν οι δικές μας μεταρρυθμίσεις. Η Πολωνία λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις ε, με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τη συνθήκη. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Ας απαντήσουμε λοιπόν σε αυτή την ερώτηση. Έχουμε την αίσθηση ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σκεφτεί και να συζητήσει όχι τι συμβαίνει στην Πολωνία, αλλά τι συμβαίνει εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σκεφτείτε γιατί επικρίνετε την Πολωνία για ρυθμίσεις που ήδη εφαρμόζονται στις δικές σας χώρες. Γιατί συζητάτε για αρμοδιότητες που η Ευρωπαϊκή Συνθήκη αναγνωρίζει στα Εθνικά Κοινοβούλια και όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλετε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συζήτηση για πολιτικά παίγνια που δεν έχουν σχέση με την κατάσταση στην Πολωνία. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη συζήτηση ως εργαλείο εκλογικής ε, μάχης σε διάφορες χώρες. Εμείς έχουμε προεκλογική εκστρατεία εν των προεδρικών εκλογών. Και μάλιστα ε, για αυτούς ε, τους λόγους ίσως ε, συζητήθηκε τώρα αυτό το θέμα για να επηρεαστεί η εκλογική διαδικασία στην Πολωνία. Σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται σε εκλογική διαδικασία χώρα μέλου. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση προ του Ευρωβουλευτέ. Μην ενδώσετε στις, ε, στην πολιτική πίεση κάποιων απογοητευμένων ε, ε, συναδέλφων που χρησιμοποιούν αυτή τη συζήτηση για τους δικούς πολιτικούς στόχους. Μερικοί πολιτικοί δεν αναγνωρίζουν ότι οι εσωτερικές πολιτικές διανέξεις όταν αναγάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εις βάρος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Η, Ευρωπαϊ... η Πολωνία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα όμως είναι μια κυρίαρχη χώρα και ως τέτοια κυρίαρχη χώρα έχει δικαίωμα και υποχρέωση να φροντίζει για τα δικαιώματα των πολιτών και της κοινωνίας της. Και η Ένωση και με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να μας αντιμετωπίσετε. Και ε, επανειλημμένως έχω πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και ως ε, Πρωθυπουργός, όταν διατέλεσα Πρωθυπουργός, σας διαβεβαίωσα ότι η πολωνική ε, κυβέρνηση τηρεί το πολωνικό σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Η Πολωνία είναι χώρα με κράτος δικαίου, αλλά είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή χώρα και κυρίαρχη χώρα. Ήταν, είναι και θα είναι τέτοια. Ευχαριστώ. εκ Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι άδικο να ακούγονται γνώμες ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή οι Ευρωβουλευτές δεν αγαπούν την Πολωνία. Είναι άδικο. Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ευκαιριακές πολιτικές σε κράτη-μέλη να καθορίζουν και να επαναδιατυπώνουν και να αλλάζουν τον οδικό χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρέχουσα κυβερνητική πολιτική στην Πολωνία έρχεται σε αντίθεση και σύγκρουση με πολλές από αυτές τις αρχές. σε θέματα κράτους δικαίου διάκριση εξουσιών ελευθερίας της έκφρασης δικαιώματα των μειονοτήτων ακόμα και στο δικαίωμα των γυναικών για έκτρωση η πολωνία και στην πολωνία από ό,τι ξέρω έχουμε κυβέρνηση. δεν έχουμε καθεστώς όχι βελτιώνονται ανανεώνονται αλλά δεν ανατρέπονται. αυτή είναι η θέση μας και σας παρακαλώ πολύ να ακούσετε όλες τις πολιτικές ομάδες και όχι την ακραία δεξιά. Ε, του EPP, το renew τους σοσιαλιστές τους πράσινους και την αριστερά. δεν είμαστε όλοι λάθος. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος ε, Πουτστεμόν ε, Κασαμάλχο ακολουθεί στη συζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα μιλάμε για το κράτος δικαίου στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Πολωνία. Είναι αναγκαίο γιατί εάν σε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τηρείται το δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο, αυτό πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με τη χώρα. Εάν το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τύχει προστασίας, τότε τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να προχωρήσουν μέχρι τέλους με κάθε κράτος, ως προς κάθε κράτος. Δεν θα πρέπει να ε, μειώνουμε τους αδύναμους και να ενισχύουμε τους δυνατούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ισπανία δυστυχώς καταστρατηγεί τα, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στην ουσία φυλακίζει πολιτικούς, καθαρά πολιτικούς ε, αντιπάλους και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική των δύο μέτρων και σταθμών. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον συνάδελφο Χαλίτσικη. Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Θα τη δεχτείτε στην αρχή. Νομίζω ότι την πήρατε πίσω. Παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα. Πραγματικά 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Κύριε Πουτσδεμόν με ε, κάθε σεβασμό. Εσείς ερχόσαστε να μας δώσετε μαθήματα για το κράτος δικαίου. Εσείς ήσασταν ο πρώτος ως πρόεδρος της ε, καταλανικής κυβέρνησης που ε, διαρρήξατε και δεν λάβατε τις αρχές και δεν τηρήσατε το δίκαιο όταν ε, στην ουσία δεν λάβατε υπόψη αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ισπανίας. Δεν θεωρείτε ότι και εσείς καταστρατηγήσατε το δίκαιο, το ισπανικό δίκαιο με τις τάσεις σας. Έτσι θα σας εξηγήσω αυτά τα δύο μέτρα και σταθμά. Αν αύριο εγώ πάω στην Πολωνία, νομίζω ότι η Πολωνία θα σεβαστεί την ασυλία μου και δεν θα με φυλακίσει. Αν αύριο το πρωί πάω στην Ισπανία, είμαι σίγουρος ότι οι Ισπανικές αρχές δεν θα αναγνωρίσουν την κοινοβουλευτική μου ασυλία. Νομίζω ότι θα με βάλουν στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής μου. Α, πρόκειται για μία στάση της Ευρώπης η οποία δεν υπερασπίζει το κράτος δικαίου εκεί που απειλείται. Ευχαριστώ. Τώρα είναι η σειρά του συναδελφού Χαλίτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Όντω, αυτή η συζήτηση δεν είναι συζήτηση για τη δικαστική μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει δικαστική μεταρρύθμιση στην Πολωνία. Ε, γιατί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι χρονοβόρα, οι διαδικασίες πανηρές. δεν υπάρχει ουσιαστική πρόσβαση των πολιτών ε, στη δικαιοσύνη. Ε, κι όμως, ε, σύμβολο των ε, τελευταίων ημερών της Πολωνίας είναι ένας, ένα μέλος της ε, κυβέρνησης που έσκησε το ψήφισμα με αλαζονικό τρόπο το ψήφισμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας που αντιτάχθηκε σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν σε τέτοια κατάσταση οι πολίτες έχουν δικαίωμα να περιμένουν ότι θα προστατευθούν τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματα του πολίτη. Και οι δικαστές είναι Ευρωπαίοι δικαστές που τηρούν το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα πρέπει να έχουμε δικαϊκές και δικονομικές εγγύσεις. Η Πολωνία δεν εκπροσωπεί η κυβέρνηση του νόμου και της δικαιοσύνης ε, δεν εκπροσωπεί τους δικαστές. Έχουμε εκατοντάδες ε, ε, δικαστές στην Πολωνία που απειλούνται από πειθαρχικές κυρώσεις λόγω της προπαγάνδας που κάνει το, η πολωνική κυβέρνηση. Και η πολωνική κοινωνία μέχρι στιγμής προστάτευσε τα δικαιώματα και τις αξίες και δεν άφησε τη καταστάσεις. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η συνάδελφος ε, Μπάρλι. Ευχαριστώ. Η ανεξάρτητη ε, ειδική της Επιτροπής της Βενετίας ε, είπαν ότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση της ε, δικαιοσύνης ε, στην Πολωνία μας έχουν φτάσει σε μια παράδεκτη κατάσταση που χρησιμοποιούνται πειθαρχικά μέτρα. Οι ειδικοί ζήτησαν να ε, σταματήσει η ψηφοφορία αυτού του νόμου, όμως φαίνεται ότι ο νόμος κυρώθηκε από τον πρόεδρο του Πολωνίας παρά τις προειδοποιήσεις. Αυτό έχει επιπτώσεις για την πολωνική κοινωνία αλλά και προσωπικές επιπτώσεις. Την περασμένη εβδομάδα το Πειθαρχικό Συμβούλιο ανέστηλε την, τον δικαστή Παύλ Σούστιτ επειδή ε, θεώρησε ότι ε, είχε ε, μιλήσει κατά ενός άλλου ε, δικαστή που είχε ήδη διοριστεί. Αυτό θεωρήθηκε λοιπόν ότι δεν ήταν σωστό. Επίσης το Πειθαρχικό Συμβούλιο θεώρησε ότι έπρεπε να προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα και με άλλους δικαστέ, το οποίο θεωρήθηκε παράνομο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έτσι, έχουμε λοιπόν πάρα πολλές περιπτώσεις. Ε, που πλέον δεν ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ε, και το Πειθαρχικό Συμβούλιο ε, παρεμβαίνει. Αυτό έχει ήδη τεθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προκειμένου να επαναφέρουμε το κράτος δικαίου. Ευχαριστούμε. Υπάρχει μια μπλε κάρτα την δέχεστε να εξηγήσω. Υπάρχουν πολλέ μόνο μία. Ε, μπορώ να δεχτώ 30 δευτερόλεπτα συνάλφο Κυριάκη. Ευχαριστώ. Εσεί είστε Γερμανίδα. Μιλάτε πολύ γενικά. Α μιλήσουμε κάτι συγκεκριμένο. Στο άρθρο 107 αναφέρονται ε, οι δυνατότητε ε, να μην ε, ε, παρακολουθούν οι δικαστικές ε, εξουσίες και απειλούνται και πειθαρχικές κυρώσεις. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Γερμανία. Κάποιος που παραβιάζει το δίκαιο μπορεί να ε, στερηθεί ως πέντε χρόνια την ελευθερία του. Οπότε ποια, ποιος νόμος είναι νόμος φήμωτρο, νόμος που φημώνει τους δικαστές, ο γερμανικός νόμος ή ο πολωνικός. 30 λεπτά, δευτερόλεπτα για την απάντηση παρακαλώ. Καταρχάς, εγώ δεν εκπροσωπώ την Γερμανία αλλά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Σίτλο επίσης ήδη ε, είπε ότι οι Γερμανοί ε, δικαστές δεν πρέπει να έχουν πολιτική δραστικαιότητα. Το AFD που είναι το αδελφό κόμμα σας ε, στην Γερμανία βρίσκεται στο Bundestag, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και το να παρακάμπτεις το νόμο είναι τελείως διαφορετικό από το να ε, ηθελημένα να παραβιάζει στον νόμο. Ε, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο το οποίο επιδικάζει υποθέσεις για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Όταν κάποιος παραβιάζει το δίκαιο, πρέπει να τιμωρείται. Δεν έχει γίνει ποτέ στη Γερμανία κάτι τέτοιο, δυστυχώ έγινε στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε στον επόμενο ομιλητή, την συνάδελφα κυρία Στρουγκάριου. Ιανουάριο δικαστές από 20 ε, κράτη-μέλη στην ουσία έδειξαν αλληλεγγύη προς τους Πολωνούς συναδέλφους. Οι Πολωνοί συνάδελφοι, οι δικαστικοί ιδιαίτερα, προσπαθούν να υπεραμεινθούν του δικαστικού του συστήματος. Αυτό που συμβαίνει στην Πολωνία δεν είναι αναθεώρηση, αλλά καταστροφή. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε αυτή την αποδόμηση σε ένα κράτος μέλος, γιατί στο νομικό μας DNA θα πρέπει, μάλλον προωθείται μέσω του νομικού μας DNA, η τήρηση του κοινοτικού δικαίου. Τώρα οι πολωνικές αρχές απομακρύνουν την χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει υπεροχή του κοινοτικού δικαίου. Μιλήσατε για αναθεώρηση. Νομίζω ότι ο Αραμπέλα ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επιστρέψτε λοιπόν στην Πολωνία και υπενθυμίστε στην Πολωνία ότι ευεργετείτε από τα κοινωνικά κοινοτικά κονδύλια και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη. Μπορεί να απαντηθεί η ερώτηση ε, αν δεχτείτε την μπλε κάρτα. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το κράτος δικαίου και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όταν είμαστε μέλη αυτού του κοινοβουλίου. η συνάδελφος Στρίκ. Με τον νόμο αυτό η Πολωνία στην ουσία ε, αποδομεί τον δικαστικό τομέα. Δεν υπάρχει ανεξαρτησία του, της ε, δικαιοδοσίας και έτσι φτάνουμε σε ένα αντιδημοκρατικό ε, κράτος, γιατί όχι μόνο δεν υπάρχουν σωστοί έλεγχοι, αλλά δεν μπορούν οι πολίτες να υπεραμεινθούν των αρχών τους κατά του κράτους. Ως προς την ατιμορρησία βλέπουμε ότι υπάρχει μία διάβρωση του κράτους δικαίου. Θα ήθελα η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει μία προσφυγή επί παραλήψη έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτό το νόμο. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το νόμο φήμοτρο και θα πρέπει να απευθυνθούμε στην πολωνική κυβέρνηση διότι υπάρχουν πολιτικές και νομικές υποχρεώσεις αλλά τώρα στην ουσία κρύβονται πίσω από την Κομισιόν. Το κράτος δικαίου έχει πυρποληθεί και πολύ σωστά οι Πολωνοί πολίτες ε, ζητούν να δράσουμε. Ε, δεχόσαστε την μπλε κάρτα από τη συνάδελφο Βυσνιέτσκα. 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η προλαλήσασα είπε ότι στην Πολωνία διαμαρτυρήθηκαν δικαστές κατά της μεταρρυθμίσει δικαστικέ οξύς και έγινε η ειρηνική διαδήλωση γιατί οι πολωνικές αρχές εξασφάλισαν την ασφάλεια των διαδηλωτών που ήρθαν από την Γαλλία και άλλες ε, πόλεις. Κάτι που δεν συνέβη στη Γαλλία με, τέτοιες, με αντίστοιχες διαδηλώσεις. Πού λοιπόν βρίσκεται η ισορροπία και η δικαιοσύνη. Ε, είναι δίκαιο να αφαιρείτε τις, ε, τις, επιδο, τις επιδοτήσεις ή τη, την περιουσία των αγροτών που όλη τους τη ζωή φρόντισαν για να μαζέψουν κάποια, κάποιο βιός και να τους, να τους ε, τα αφαιρείτε έτσι αμέσως. Είναι δικαιοσύνη αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτή η ερώτηση. Αναφερθήκατε στον προλαλήσαντα, ο οποίος μίλησε για μία ειρηνική διαδήλωση, γιατί ακριβώς ε, ζητήθηκε να μην φημώνονται οι δικαστές και να μπορούν να κρίνουν αβίαστα και ανεξάρτητα. Η δημοκρατία σημαίνει ότι προστατεύουμε τους πάντες και τις μειονότητες και η δημοκρατία και το κράτος δικαίου κινούνται χέρι-χέρι. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ο συνάδελφος Κοζάν Λεσπόνς έχει το λόγο. Οι πολωνικές αρχές ε, ενδιαφέρονται περισσότερο στην αντιπαλότητα παρά στη συμμόρφωση. Η Επίτροπος Γιούροβα ζήτησε να υπάρχει ένας σωστός και διαφανής διάλογος. Ε, δυστυχώς στη συνέχεια πάλι έγινε επίθεση στο δικαστικό τομέα. Από τον Ιανουάριο έχουν μπει 40 δικαστές στο στόχαστρο διότι δεν δέχονται τις αποφάσεις του, της κυβέρνησης τι δικαιοσύνη υπάρχει όταν διώκονται οι δικαστές, τι θέλουμε να ε, βελτιώσουμε τον δικαστικό τομέα ή να χειραγωγείται ο δικαστικός τομέας από το κράτος. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Αυτό που βλέπουμε στην Πολωνία ε, δεν είναι αναθεώρηση αλλά καταστολή. Όταν ε, τίθεται εν κινδύνο το δικαστικό σώμα, τότε θα πρέπει να παρέμβουμε και εμείς, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έτσι ώστε να τηρηθεί το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και άλλη μπλε κάρτα. Να σας εξηγήσω όμως ότι ο κανονισμός προβλέπει μόνο μία μπλε κάρτα ανομιλητή. Οπότε, κυρία Βυσνιεύσκα, εσεί μιλήσατε με τη διαδικασία τη μπλε κάρτα. Άμα θέλει κάποιο άλλο να υποβάλει ερώτηση με μπλε κάρτα, πολύ ευχαρίστω να τη δέχεται ο μιλητή. Αλλά όχι δεύτερη μπλε κάρτα από τον ίδιο άνθρωπο, από την κυρία Βυσνιεύσκα, ε, προκειμένου. Ο κύριο Μπιέντρον. Από την ανάληψη τη εξουσία από το νόμο και δικαιοσύνη, ο Υπουργό Δικαιοσύνη και Γενικό Αγγελέα Σμπίκινε Ζόμπρο ε, προσπαθεί να καταστρέψει το πολωνικό δικαστικό σύστημα. Έχει συνεχεί τριβέ και αντιπαράθεση και με του ε, Πολωνού πολίτε και με το θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολωνική κυβέρνηση θέλει να περάσει την επόμενη καταστροφή, να παγώσουν τα κοινοτικά κονδύλια προ την Πολωνία και σιγά σιγά να οδεύσει προς, προς μια αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς ένα πολέξιτ και όλα αυτά για να προστατεύσει τα κομματικά συμφέροντα. Αυτές είναι οι πραγματικές απειλές που δυστυχώς τα σπασμένα θα τα πληρώσουν οι απλοί πολίτες της Πολωνίας. Ε, ακόμη δυστυχώς στην Πολωνία δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των πολιτών, παρά μόνο εφόσον ε, είναι μέλη του κυβερνώντος κόμματος. Αν θέλει η Πολωνία να γίνει κράτος δικαίου θα πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση. Γιατί σήμερα μιλούμε για το κράτος δικαίου και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τους απλούς πολίτες που μερικές φορές λόγω της ανικανότητας και της α, ε, α, ε, παραφροσύνης της ε, πολωνικής κυβέρνησης θα πληρώσουν τα σπασμένα, θα είναι τα θύματα αυτής της κατάστασης και θα οδηγηθούν λόγω της δικής σας παραφροσύνης προς ένα πολέξιτ, προς μια αποχώρηση Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μπλε κάρτα, ε, κύριε Μπέντρον, για σας. Τη δέχεστε. Ναι, η κυρία Ξαφτσίνσκα. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, όποιος μιλάει για το Polexit θέλει απλώς προβλήματα και σκάνδαλα. Είμαι ευρωβουλευτής που εξελέγει στην Πολωνία. Είμαι Πολωνέζα, και περήφανη για τη χώρα μου, για την πατρίδα μου και την ιστορία μου. Μη φοβίζετε τον κόσμο με το πολέξιτ, Ε, δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Έχετε μισό λεπτό για την απάντηση, κύριε Μπέντρον. Κυρία συνάδελφε, και εγώ είμαι υπερήφανος για την πατρίδα μου. Είμαστε η χώρα που έχουμε το αρχαιότερο σύνταγμα. Είμαστε χώρα που ανέτρεψε τον κομμουνισμό. Είμαι περήφανος για αυτά. Ντρέπομαι όμως που στην πατρίδα μου υπάρχουν άνθρωποι που είναι χειρότεροι από τους κομμουνιστές, που προσπαθούν να καταστρέψουν τη χώρα ακόμη περισσότερο από ό,τι οι κομμουνιστές. Αυτό είναι ντροπή για τη σημερινή κατάσταση στην Πολωνία. Παρακαλώ, όχι εσωτερική συζήτηση. Δεν επιτρέπεται συζήτηση. Ε, αλλά μόνο υποβολή ερωτήσεων με την μπλε κάρτα. Εσείς δεν κάνατε καμία ερώτηση με την μπλε κάρτα. Στην επόμενη ε, μπλε κάρτα θα ήθελα παρακαλώ να υποβληθεί ερώτηση και να μην χρησιμοποιείτε τη διαδικασία αυτή για να έχετε επιπλέον χρόνο αγόρευση. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Ζούροβα, κύριε Άντερς, ε, και Αγαπητέ Προεδρεύοντα, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για γεγονότα του Γκτάνσκ. Τα γεγονότα του Γκτάνσκ οδήγησαν στα, στις 27 σημαίες μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σεβόμαστε τους Πολωνούς, όμως δεν τους αναγνωρίζουμε μέσω της κυβέρνησης αυτή η πειθαρχική διαδικασία ε, και η δίθεν αναθεώρηση του δικαστικού τομέα είναι απαράδεκτη. Δυστυχώς υπάρχει πλήρης αποδόμηση ενός ιστορικού και εκτιμένου. Πρόκειται για έναν προμαχώνα, τον προμαχώνα του κράτους δικαίου, τον οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το χώρο των ελευθεριών και της δικαιοσύνης για να προωθήσουμε φιλόδεξα σχέδια, για να μην δεχτούμε την, τρομοκ, την επιγραμμική τρομοκρατία. Ποιες δράσεις θα προβάλλετε για να δοθεί τέλος σε αυτή την κατάσταση που οδηγεί, σε μια ευάλωτη Ευρώπη ως προς το κράτος δικαίου. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τον συνάδελφο Μπίλτσενγκ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε Γιούροβα, Είμαι ένας ε, περήφανος Ευρωπαίος από, μια, από την Κεντρική Ευρώπη. Πριν από 30 χρόνια αποφασίσαμε δημοκρατικά να επιστρέψουμε σε μια δημοκρατική και ελεύθερη Ευρώπη. Αυτή η επιστροφή άλλαξε θεμελιωδώς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το καλύτερο, η ειρήνη και η δημοκρατία απλώθηκαν στην Ήπειρο. Υπάρχει η ευρωπαϊκή αξιοπρέπεια, η αφοσίωση στους κανόνες, τη δικαιοσύνη, όλα αυτά τα βλέπουμε σε όλες τις γωνιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Σοβλοβάκος ανησυχώ όμως για την ποιότητα της δικαιοσύνης και την αξιοπιστία των κανόνων σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό εδώ θέλω να περασπιστώ και την πολωνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Πιστέψτε με, πραγματικά δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα. Ε, πέραν από την ανησυχία μας για την ποιότητα της δημοκρατίας και την ποιότητα του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Προς όφελος λοιπόν όλων των Ευρωπαίων δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την επιστροφή της κατάχρησης της δικαιοσύνης στην Ευρώπη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον συνάδελφο Μάντλ. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε το γεγονός ότι έχουμε στενές σχέσεις ε, και συναισθανόμαστε τους πολίτες ε, στην Πολωνία ως Αυστριακός, Η Αυστριακοί έχουμε ε, πολλά να οφείλουμε ιστορικά στην Πολωνία. Η ιδεολογία του 20ου αιώνα έπρεπε δυστυχώς ε, υπέφερε πολλά. Ε, άρχισε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την επίθεση στην Πολωνία. Τα εθνικοσοσιαλιστικά εγκλήματα εκεί ε, ξεκίνησαν και ταυτόχρονα να πω ότι οι Πολωνοί αυτή την ηγεσία που θέτει υπό αμφισβήτηση το κράτος δικαίου δεν την αξίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέλουν, πρέπει και αξίζουν να ζουν σε ένα κράτος δικαίου με ένα δίκαιο μέλλον για τα παιδιά τους. Ένα κράτος δικαίου που το έχουν κερδίσει. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον ε, συνάδελφο Μουρεζάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Πολωνίας ε, και το κόμμα του νόμου και της δικαιοσύνης λέει ότι τηρεί το κράτος δικαίου αλλά δρά κατά του κράτους δικαίου καθημερινά. Θα πρέπει να δούμε τις δράσεις αυτής της κυβέρνησης και όχι τις δηλώσεις της. Αυτό που λέει ε, στην λαό της η κυβέρνηση της Πολωνίας μέσα από αυτή την μεταρρύθμιση απόφαση του δικαστικού σώματος ε, είναι στην ουσία κάτι που αυτοί αποκαλούν αποκομμουνιστικοποίηση, όμως ε, είναι απολυταρχία. Εμείς ε, γνωρίζουμε ότι η Πολωνία είναι κάτι παραπάνω από ότι είναι η τρέχουσα κυβέρνησή της. Οι κυβερνήσεις πάνε και έρχονται. Είναι μια χώρα που προστατεύει την ανεξαρτησία των δικαστών και το κράτος δικαίου ε, παρά ε, ε, τον εκφοβισμό. Είναι μια χώρα που είναι πεισμένη για το κράτος δικαίου, που έχει αντικειμενική δημοσιογραφία, που προωθεί την ελευθερία του λόγου, αψηφώντας την πολιτική προπαγάνδα. Είμαστε λοιπόν στο πλευρό του πολωνικού λαού και λέμε στην πολωνική κυβέρνηση να ακούσει τη φωνή του λαού της. Ευχαριστούμε. Υπάρχει μια μία μπλε κάρτα από τη συνάδελφο Ξαλεύσκα. Την δέχεστε. Μισό λεπτό για ερώτηση, ερώτηση. Αν όχι θα διακόψω. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, αλλά... Ε, 20.000 ε, ε 20.000 ε, πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους στηρίζοντας ε, τα μέτρα της πολωνικής κυβέρνησης. Το έχετε υπόψη. Επίσης, ε, σε καμία διάταξη της Ευρωπαϊκής Συνθήκης δεν αναφέρεται αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεξαγωγή τέτοιων συζητήσεων. Επίσης, κυρία Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να επιτρέπετε τη χρήση επιθέτων εις βάρος κάποιας χώρας. Δεν θα πρέπει να προσβάλλουμε ή να βρίζουμε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πού είναι η ερώτησή σας. Γιατί η μπλε κάρτα προϋποθέτει ερώτηση για να απαντήσει ο συνάδελφος. Τελευταία φορά ήταν που έδωσα μπλε κάρτα, γιατί η μπλε κάρτα είναι για ερώτηση, όχι για να παρατείνετε το χρόνο ομιλία σας. Μισό λεπτό, αλλά μόνο για υποβολή ερωτήσεων είναι οι μπλε κάρτες. Η ερώτηση ήταν σαφής. Κατά πόσο γνωρίζω τη συνθήκη των της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνθήκη περί λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω πολύ καλά τις συνθήκες καθώς και τα άρθρα που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές αξίες και θα πρέπει να υπερασπιστούμε το κράτος δικαίου σε κάθε γωνιά της Ευρώπης γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες. Ξέρω για τις δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στην Πολωνία που ε, καταφέρθηκαν κατά της κυβέρνησης και εμείς είμαστε αλληλέγγυοι με αυτούς. Προχωρούμε στη σειρά. Ο επόμενος είναι ο συνάδελφος ε, Ποσπίλσιλ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Σίντουο Αναφέρθηκε στην ομιλία τη στην Τσεχία, στην Δημοκρατία της Τσεχίας. Για πέντε χρόνια διατέλεσα υπουργό δικαιοσύνη στην Τσεχία και πουδενή, ουδέποτε δεν ε, διώξαμε δικαστές στην Τσεχία. Μπορεί να επιβάλλονται κάποιε πειθαρχικέ κυρώσει σε δικαστέ για καθυστερήσει ε, των ε, δικών, αλλά ουδέποτε δεν επιβάλαμε κυρώσει σε δικαστέ για τι απόψει του, για τη γνώμη του. Η μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσία στην Πολωνία δεν έχει καμία σχέση με οποιασδήποτε δικαστικές μεταρρυθμίσεις έγιναν στη Τσεχία. Και δυστυχώς δεν θέλετε συμβαστική λύση ή συνεργασία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σας ήδη υπέγραψε το νόμο αυτό. Ε, δεν θα πρέπει να ποινικοποιείτε οι δικαστές για την έκφραση της γνώμη του. Μόνο ε, όταν καθυστερούν οι δίκες μπορούν να επιβάλλονται πειθαρχικέ κυρώσεις στις δικαστές, όχι όμως για έκφραση προσωπικών απόψεων όπως κάνετε εσείς. Ευχαριστώ. Κύριο Σικόρσκι. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώ. Στην Πολωνία καταστρατηγήθηκε το κράτος της ε, Πολωνίας ε, κατηγόρησε τον Ντόναλτ Τούσκ για ε, μη καλή διαλεύκανση της, ε, του αεροπορικού ατυχήματος του Σμόλεσκ. Και μάλιστα κατηγορήθηκε επανειλημμένος από την ε, πολωνική κυβέρνηση ο Ντόναλτ Τούσκ. Και μάλιστα σήμερα με, την, με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης ασκήθηκε δίωξη κατά του Τούσκα παρόλο που ο, ε, ο κύριος Τούσκ ισχυρίζεται ότι είναι αθώος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη λοιπόν στην Πολωνία. Παρακαλώ την Επίτροπο Γιώροβα να κάνει ό,τι μπορεί για να επανέλθει το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Έχω πολλές αιτήσει για κάτι Δυστυχώ δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλους του συναδέλφους. Θα επιτρέψω έναν ομιλητή ανά ομάδα και όχι σε όσους ήδη έχουν λάβει μέρο στη συζήτηση μέχρι στιγμής. Ξεκινάμε με τον κύριο Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κοινοί κανόνες και αξίες και εάν τίθενται σε κίνδυνο τότε θα πρέπει να αντιδράσουμε. Η κατάσταση είναι απόλυτα σαφής. Δυστυχώς δεν τηρείται το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος και γι' αυτό δεν υπάρχει και αμοιβαία εμπιστοσύνη με το κράτος αυτό. Θα ήθελα η κυρία Σέντλο να θυμηθεί όταν ήταν Πρωθυπουργό, ότι μιλήσαμε για συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησής της και μας είπε ότι θα δεχτεί τα αποτελέσματα της Επιτροπής της Βενετίας. Τίποτα τέτοιο δυστυχώς δεν συνέβη και σήμερα μας λέτε ότι οι δικές σας μεταρρυθμίσεις πήγαν πολύ καλά. Θα έπρεπε να ντρέπεστε γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Σπούρεκ. Ευχαριστώ. Εξαπλάγιν, όταν μετά από συζήτηση με την Ursula von der μου είπε ότι ε, αντικείμενο της συζήτηση δεν ήταν το κράτος δικαίου. Πώς είναι δυνατό η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συναντήσει τον Πολωνό Πρωθυπουργό και να μην συζητήσουν το κράτος δικαίου. Η Κροατική Προεδρία δυστυχώς δήλωσε ότι δεν είναι προτεραιότητά της ε, το κράτος δικαίου. Και όμως εμείς έχουμε συνεχείς συζητήσεις για το κράτος δικαίου και ξέρουμε πόσο αναποτελεσματικές είναι κάποιες δράσεις, πόσο αναποτελεσματικό είναι το άρθρο 7. ακόμη και η αιρεσιμότητα δεν εφαρμόζεται για την αναστολή των κοινοτικών κονδύλιων. Θα πρέπει ε, να μην πλήξουμε τους πολίτες και θα φροντίσουμε γι' αυτό. Και νομίζω ότι ο καιρός της διπλωματίας έχει περάσει. Περιμένουμε από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφείς δηλώσεις και δράσεις. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους Πολωνούς πολίτες και τους Πολωνούς δικαστές που προστατεύουν το Πολωνικό Σύνταγμα. Περιμένουμε συγκεκριμένες δράσεις, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιώβεβα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου. Το Κοινοβούλιο το 2017 επανέλαβε ε, πολλές φορές ότι η κατάσταση στην Πολωνία ε, θίγει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εμείς διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση αυτή ισχύει από το 2016 και εξής. Τίποτα όμως δεν βελτιώθηκε, γιατί με αυτή τη μεταρρύθμιση μπορούν να απολυθούν δικαστές και έχει επιδεινωθεί η άρδινη κατάσταση. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να παγώσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια προς την Πολωνία ή να καταβάλλονται υπό συνθήκες, δηλαδή μόνο αν βελτιωθεί η κατάσταση, τότε μόνο να καταβαλλονται υποσυνθηκες να χορηγείται η χρηματοδότηση αυτή. Η παράβαση των κανόνων θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κάθε φορά που είμαστε στο Στρασβούργο, λέω ο Σάλφος συζητάμε για την κατάσταση στην Πολωνία πραγματικά. Ε, με τι ζήλο η Πολωνία από τα αριστερά και το κέντρο ε, επιτίθενται ε, στην ε, πατρίδα τους. Έχουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης Νοεμβρίου επειδή οι, δεν, αναφε, δεν διορίζονται οι δικαστές από το δικό του συμβούλιο αλλά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ε, δίνεται ε, μία τέτοια απόφαση ε, και αυτό που ζητάτε από την Πολωνία δηλαδή οι ίδιοι δικαστές να διορίζουν το, τους ομοίους τους είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το διαχωρισμό των εξουσιών, δηλαδή ανεξαρτησία των αποφάσεων, τον διορισμό, αλλά όχι διορισμό του ιδίου ε, του συναδέλφου μας. Συνεχίζουμε με τον συνάδελφο Τόμασιτς. Τη συνάδελφο Τόμασιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Πολωνία βρέθηκε στο στόχαστρο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων γιατί θέλει να εκδημοκρατήσει το πολιτικό και δικαστικό τη σύστημα. Αυτό είναι η θλιβερή αλήθεια που θα πρέπει να την κοιτάξουμε κατάματα. Ε, γιατί η έλλειψη κατανόηση που δείχνει η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Πολωνίας οδηγεί σε διένεξη που δεν είναι προς το συμφέρον κα, κανενός. Θα πρέπει οι παλιές δημοκρατίες να καταλάβουν ότι οι πιο νέες χώρες ε, ε, οι πιο νέες δημοκρατίες δεν μπορούν να φτάσουν τόσο γρήγορα στις δικές τους προδιαγραφές. Έχουμε λοιπόν ουσιαστική διαφορά και οι χώρες που επιβίωσαν από το παλιό κομμουνιστικό σύστημα και καθεστώς και μετατράπηκαν σε δημοκρατίες ε, προσπαθούν ε, να κάνουν μία μετάβαση και να εξαρθρώσουν το παλιό κομμουνιστικό τους παρελθόν. Επιτρέψτε μας αυτή τη μετάβαση που χρειαζόμαστε όλες οι χώρες που περάσαμε από το κομμουνιστικό καθεστώς. Θα ήθελα να σα κάνω μια εξήγηση, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί βλέπω και νευρισμό. Δήλωσα από την αρχή ότι θα επιτρέψω μόνο έναν ομιλητή ανά πολιτική ομάδα για το Catch Η δική σα ομάδα είχε, είχε, είχε ήδη εκπροσωπηθεί το ECR. Περνάμε τώρα στι τελικέ παρεμβάσει. Ο Επίτροπο Ρέντερ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητά μέλη. Επιτρέψτε μου να επανέλθω σε ορισμένα ζητήματα που εθίγησαν κατά τη συζήτηση ως προς το νέο νόμο, γιατί πράγματι από την προηγούμενη συζήτηση, ορισμένες εβδομάδες πριν, ανέκυψε νέος νόμος. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε έναν ε, δίκαιο διάλογο με όλα τα κράτη-μέλη για να επανορθωθεί η κατάσταση, αλλά δεν θα οροδίσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα όταν υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με ένα νόμο. Υπάρχουν λοιπόν ανησυχίες ως προς τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο, γιατί φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου καθώς και η ανεξαρτησία του δικαιοδοτικού και δεν υπάρχει, δεν τηρείται το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ως προσχόλια ορισμένων μελών θα ήθελα να επαναλάβω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η εργάνωση του δικαιοδοτικού εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, αλλά κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος και καθήκοντος, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με βάση τις υποχρεώσεις δυνάμει του κοινοτικού δικαίου, το οποίο σημαίνει τήρηση του κράτους δικαίου, ιδιαίτερα την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, διότι τα πολωνικά δικαστήρια είναι ευρωπαϊκά δικαστήρια και γι' αυτό οι πολωνοί πολίτες θα πρέπει να ευεργετηθούν από τα δικαιώματα που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο. Γι' αυτό ανησυχώ για τον, ως προς τον νέο αυτό νόμο και θα ήθελα να σας τονίσω ότι η Επιτροπή είναι θεματοφύλακας των συνθήκων και μέσα στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου δικαιοσύνης θα λάβω κάθε μέτρο που χρειαστεί. Το πειθαρχικό τμήμα συνεχίζει να λειτουργεί παρά τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά τις αποφάσεις της 19ης Νοεμβρίου. Το πειθαρχικό λοιπόν τμήμα δεν αποτελεί δικαστήριο δυνάμει του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου. Θα ήθελα να πω ότι οι ε, αποφάσεις ερμηνείας του δικαίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να τηρούνται πλήρως και τα κρατικά δικαστήρια θα πρέπει να δέχονται την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στις 4 Φεβρουαρίου του 2020 ε, στην ουσία ε, ανέστηλε τη λειτουργία, μάλλον έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν δικαστή ο οποίος δεν δέχτηκε την απόφαση του Πολωνικού Δικαστηρίου με ε, φυσικά μείωση του, της αμοιβή του. Οπωσδήποτε τα δικαστήρια αποτελούν μία ανεξάρτητη αρχή. Δυστυχώς όμως το πειθαρχικό τμήμα λειτουργεί. Επέλεξε έξι υποψηφίους δύο εκ των οποίων είναι μέλη του Εθνικού Δικαιοδοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε σχέση με το Συνταγματικό Δικαστήριο ότι η δυνάμει της πρότασης του Δεκεμβρίου που ε, επικαλείται το άρθρο 7 της συνθήκης δυστυχώς ε, υποσκάπτονται οι αποφάσεις των πολωνικών δικαστηρίων και η συνταγματικότητά τους. Υπ' αυτή την έννοια, μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, χρειάστηκε να γίνουν νέες προσφυγές. Πολλές φορές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάσταση οδηγεί σε ένα δικαστικό χάος. Η επανόρθωση θα σήμαινε ότι τηρείται η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εργάζεται σε σχέση με τη δημιουργία ενός προληπτικού μηχανισμού λειτουργίας του ε, δικαιοδοτικού τομέα σε σχέση με τις διάφορες ερμηνείες του κράτους δικαίου. Θα βασιστούμε σε συγκεκριμένες πηγές για να δούμε πώς έχει η επιτόπια πραγματικότητα. Έτσι θα μπορέσουμε να, ε, μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε ζητήματα ερμηνείας του κράτους δικαίου και θα καλύπτονται όλα τα ε, κράτη-μέλη ομοίως. Η πρώτη έκθεση για το κράτος δικαίου ε, βρίσκεται σε μία φάση κατάρτισης και είμαστε σε επαφή με ένα συγκεκριμένο δίκτυο για την ερμηνεία του κρατικού δικαίου με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα ήθελα να είμαι σαφής και να πω ότι αυτός ο μηχανισμός ε, δεν αντικαθιστά τη διαδικασία επί παραβάση ή το άρθρο 7 εκεί που χρειάζονται. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανόμενης και της Πολωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο και τώρα συνεχίζουμε με την ε, κυρία ε, Υπουργό, την κυρία Μπρίνιετς. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η Προεδρία και το Συμβούλιο συνολικά αποδίδουν μεγάλη σημασία στο κράτος δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι στην καρδιά των προσπαθειών μας και θα λάβουμε υπόψη μας τις απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα στη συζήτηση όσον αφορά τα επόμενα βήματα στο άρθρο για το άρθρο 7 στο Συμβούλιο παρόλο που το κράτος δικαίου είναι ε, μία από τις προτεραιότητες ε, της Κροατικής Προεδρίας ε, δεν μπορούμε να κρίνουμε τις, την έκβαση της διαδικασίας παρακολουθούμε στενά τα εξελίξεις και θα δούμε τι θα γίνει στο στην επόμενη συνάντηση του, Υπουργείου... του της Επιτροπής Γενικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Και εδώ κλείνει η συζήτηση. Πριν ε, πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ε, να σας πω ότι σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 28 Ιουνίου του 2018 και τον Ιανουάριο του 2020, στις 31 Ιανουαρίου 2020, ε, φεύγει ε, το Ηνωμένο ε, Βασιλείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κρότσος, η κυρία Ντορμάκεν και ο κύριος Μάσελ Τεγκράφ